Ε, περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα που είναι μια κοινή συζήτηση για τους αναπληρωτές δικαστές. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια έκθεση της κυρίας Στάιν που αφορά τους αναπληρωτές δικαστές. Επίσης και μια έκθεση επίσης της κυρίας Στάιν που αφορά το πρωτόκολλο σχετικά με τον οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταρχάς να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια η κυρία Τάιν, παρακαλώ. Κύριε Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε. Άσε. Κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο έχει υπερβαλλικά πολλή εργασία. Αυτό που θα αποφασίσουμε αύριο μπορεί να έχει τεχνική φύση από πρώτη άποψη. Αφορά το νέο οργανισμό των τριών δικαστηρίων. Από τα οποία αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά από πίσω υπάρχουν περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες ε, μέσω τελευταία και της συνθήκης Λισαβόνας. Οπότε και οι αρμοδιότητες του δικαστηρίου έχουν ε, βαθμιαία αυξηθεί. Η υπερφόρτωση εργασίας, ο, υπερβολικό, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας δεν έχει να κάνει με τόσο πολλές νέες περιπτώσεις, αλλά με το γεγονός ότι έχουν ε, εισαχθεί 12 νέα κράτη-μέλη. Οπότε υπάρχουν νέα τμήματα δικαίου. Και γι' αυτό υπάρχουν μεγάλε επιπτώσει από τον τρόπο λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για τον τρόπο λειτουργία τη Ένωση και για την ζωή των πολιτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν συμμετάσχει στον τριμερή διάλογο από την αρχή να συνεργαστούν και να βρούμε του σωστού συμβασμούς. Αυτό εν μέρη το επιτύχαμε. Θα αρχίσω με το τμήμα όπου επιτύχαμε του σωστού συμβασμού για να υπάρξει καλύτερη λειτουργία του δικαστηρίου και καλύτερη διαδικασία. Είναι τα εξή σημεία με πρόταση του ίδιου του δικαστηρίου θα δημιουργηθεί ο θεσμός ενός αντιπροέδρου που θα μπορεί να βοηθήσει τον πρόεδρο για τις διοικητικές υποθέσεις και θα συμμετέχει και στις ολομέλειες. Επίσης, ε, το κύριο σώμα θα αποτελείται από 15 ε, δικαστές, ούτως ώστε θα γίνει και καλύτερη κατανομή της εργασίας και οι προτάσεις για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης είναι ε, επίσης θετικές. Θα αποτελείται αυτό το δικαστήριο από 7 δικαστές. Και επειδή είναι τόσο λίγοι δικαστές, εάν έστω ένας και μόνο είναι άρρωστος, ε, περιορίζεται πολύ η δυνατότητα δράσης. Γι' αυτό θέλουμε να ορίσουμε αναπληρωτές δικαστές θα γίνεται ο ορισμός τους με κάποια σειρά, με βάση ένα κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο, εάν κάποιος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, θα μπορούν να πάρουν τη θέση του. Αυτή είναι η σωστή συμβασμή με τους οποίους επιτύχαμε και για τους οποίους ευχαριστώ όλους τους εμπλεκομένους. Αλλά όπως είπα δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για όλα τα θέματα. Αυτό έχει να κάνει και θέλω να το τονίσω όχι μόνο ε, με ευθύνη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, αλλά με ορισμένε εθνικές αρχές κάποιων κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα, ζητήθηκε να ανέβουν στους 39 δικαστές από 27. Αυτό βεβαίως είναι σωστή διαδικασία, γιατί ε, βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε για το πόσοι ακριβώς πρέπει να συμμετάσχουν. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η αύξηση του αριθμού των δικαστών θα βοηθήσει σε καλύτερη δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να παίζει ε, ουσιαστικό ρόλο από ποιο κράτο μέλο προέρχονται οι επιπλέον δικαστέ, αλλά μόνο τα προσόντα του, Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει η αρχή τη ανεξαρτησία των δικαστών. Αλλά αυτά είναι για το μέλλον. Έχουμε προτείνει επανειλημμένα διάφορε διαδικασίε για να ορίζουμε σωστά του δικαστέ, Αλλά τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο δεν δέχτηκαν καμία από αυτέ τι λύσει. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα αποφασιστεί αύξηση του αριθμού των δικαστών στο εγγύ μέλλον αυτά τα θέματα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με εθνικές ε, προκαταλήψεις. Είναι πολύ μη ικανοποιητική κατάσταση. Στο μέλλον πρέπει να φροντίσουμε το ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται ε, σε εύλογο χρόνο. Εάν αργούν πολλοί οι αποφάσεις, μέχρι και 5,5 χρόνια, αυτό είναι παραβίαση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο τα κράτη-μέλη, λόγω των εξαιρετικά αντικειμενικών προτάσεων, να αποφασίσουν επιτέλους για να μην μειωθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς. Ευχαριστώ κυρία Τάιν. Άλλοι ομιλητέ τώρα, πέντε λεπτά. Ο κύριος Μαυρογιάννης, από πλευράς του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο που αποφάσισε να διεξαγάγει αυτή την κοινή συζήτηση για τις δύο εκθέσεις της κυρίας ε, Τάιν για τις προτινόμενες τροπολογίες στον οργανισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το σχέδιο κανονισμού που αφορά αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επικοδομητική και θετική αντιμετώπιση της για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Επίσης θέλω να αποτίσω φορό τιμής και στη Δανέζικη Προεδρία που έπαιξε ουσιαστικό ρόλο για να σημειωθεί ταχεία πρόοδος εντός του Συμβουλίου καθώς και στη συζητήση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η καλή συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το σημαντικό θέμα έχει οδηγήσει σε ταχεία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα όντω. Στόχος αυτών των δύο προτάσεων είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνολικά και ιδιαίτερα να επιτρέψει το δικαστήριο να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο όγκο υποθέσεων και ε, το σημαντικό αριθμό υποθέσεων που καθυστερούν. Θέλουμε να υπάρχει νομική βεβαιότητα και αποδοτικότητα. Έχω πλήρη συνείδηση ότι χρειάζεται περαιτέρω εργασία σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά την αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, και τα δύο θεσμικά μας όργανα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν ούτω ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. Να στραφώ τώρα στα διάφορα στοιχεία του ε, συμβαστικού πακέτου επί του οποίου θα ψηφίσετε αύριο θα υποβάλουμε μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας των τριών δικαστηρίων που αποτελούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα τελευταία χρόνια το δικαστήριο έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές και όσον αφορά τον όγκο αλλά και τη φύση των υποθέσεων. Αυτό οφείλεται και σε εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο σε διάφορους τομείς και στη διεύρυνση της Ένωσης. Τα μέτρα που περιέχονται στα κείμενα που έχετε ενώπιόν σας θα επιτρέψουν στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ένδικες διαδικασίες και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία στοιχεία. Πρώτον, η δημιουργία του θεσμού του Αντιπροέδρου και στο Πρωτοδικείο και στο ε, Γενικό Δικαστήριο. Θα βοηθήσουν τους Προέδρους στις αρμοδιότητές τους. Δεύτερον, η αλλαγή της σύστασης ε, του διευρουμένου δικαστηρίου και η δυνατότητα να υπάρχουν αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης για να αναπληρώνουν δικαστές που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν για λόγους υγείας στις ένδικες διαδικασίες. Τα άλλα στοιχεία της πρότασης που έχουν να κάνουν με την αύξηση του αριθμού δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο σας διαβεβαιώ ότι το Συμβούλιο έχει πλήρη συνείδηση της ανάγκης να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα επιγόντως. Ωστόσο, είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα αυτό εντός του Συμβουλίου. Η Κυπριακή Προεδρία είναι αποφασισμένη να βρει λύση. Αλλά θα το κάνουμε αυτό με τρόπο ώστε να λαμβάνει πλήρως υπόψη την πλήρη γάμα απόψεων εντός του Συμβουλίου. Χαίρομαι που μπορούμε να προσβλέψουμε να προσβλέπουμε στην έγκριση των δύο προτάσεων αυτών που συζητάμε σήμερα το απόγευμα. Προσβλέπω στη συνέχιση της θαυμάσιας συνεργασίας με το δικαστήριο για τα θέματα που ακόμη είναι προς και είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε νωρίς σε αποδεκτή λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μάλστρον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επικοδομητική της στάση. Λυπάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η απόφαση για επιπλέον δίκαστες αναβάλλεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. παρόλα αυτά, η συμβιβαστική λύση στην οποία έφτασαν τα διάφορα όργανα σήμερα είναι κάτι το θετικό. Κάποιες από τις αλλαγές τις οποίες είχαμε προτείνει τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η πρόθεση του Κοινοβουλίου να διοργανώσει μια συζήτηση ε, για την ουσία σχετικά με τις, διαφορετικέ τις διαφορετικές απόψεις πριν από την δημοσίευση της απόφασης είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην επικοδομητική εξέλιξη των συζητήσεων. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω την κυρία Βέρτμαν. Δεν είναι σε αυτή τη φάση εδώ. Το ίδιο ισχύει επίσης και με τον κύριο Μέστερσμιτ, ούτε και αυτός είναι εδώ. Και μπορούμε να περάσουμε αμέσως στον κατάλογο των ομιλητών. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για δύο λεπτά ζύφκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να είναι ένα σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση της ευρύτερης της προβληματικής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος. Η συζήτηση τώρα ξεκινάει και θα γεννήσει στο μέλλον πολλές επιμέρους συζητήσεις. Σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασιζόμενη σε αυτήν, περιμέναμε κάτι περισσότερο. Δεν πιστεύαμε ότι η διαδικασία θα ήταν τόσο δύσκολη και δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν τόσες διαφορές ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Οι προσωρινοί δικαστές για το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει τη λειτουργία του δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά το βασικό συστατικό της μεταρρύθμισης αυτής είναι η απόφαση για την αύξηση των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται ποτέ κάποιες ε, προτάσεις αλλαγών οι οποίες από κάποιους θεωρούνται ρηξικέλευτες. αλλά παρόλα αυτά είναι σαφές ότι το θέμα θα πρέπει να έρθει προς συζήτηση εκ νέου του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις συνθήκες, οι οποίες όμως μερικές φορές είναι ιδιαίτερο χρονοβόρες και αυτό δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες μας. Μάλιστα τώρα θα υπάρξει και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κροατία θα γίνει σύντομα μέλος. Θα, ενταχθεί και στην, θα ενταχθούμε και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αυτό σημαίνει περισσότερη ύλη για τα δικαστήρια. Νομίζω ότι τα δικαστήρια μας χρειάζονται νέα νομικά μέσα και τους πόρους, τους ανθρώπινους που θα τους επιτρέπουν να καλύψουν τις νέες ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στην απονομή δικαίου. Ταυτόχρονα Οι χρονοβόρες διαδικασίες προκαλούν ιδιαίτερα υψηλές ζημίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά. κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αναπρωτήπου και κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την επικοδομητική εργασία που επετέλεσε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει συνεχώς υπερβολικό φόρτο εργασίας. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η Ένωση διευρύνθηκε με 12 κράτη-μέλη και επίσης ε, διευρύνθηκαν και αρμοδιότητές της. Άλλαξε λοιπόν ο κανονισμός ούτω ώστε σε θέματα όπως η πνευματική ιδιοκτησία να μπορεί να αποφεύγεται η ακροματική διαδικασία. Οι πολίτες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ε, απέτηση να αποφασίζεται σωστά και έγκαιρα. Και μπορεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου να αποστέλει σε τμήματα ε, ορισμένα θέματα. Από αυτές τις ε, διάφορες προτάσεις που έχουν, που έχουν γίνει επελέγει καλύτερη. Άλλαξε λοιπόν ο κανονισμός ε, με βάση και τις ηθίκες Λισαβόνας. Με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ελαστικότητα γιατί η κατάσταση είναι επίγουσα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρέπει να ε, αποκτήσει 39 δικαστές. Αυτή είναι η γνώμη και του εισηγητού. Όμως θα ήθελα να ξέρω με ποια κριτήρια κατέληξε σε αυτόν αριθμό, τον, ε, ακριβώς τον αριθμό. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά δέχομαι τον αριθμό. Βεβαίω, ε, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για τους δικαστές. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να είναι και καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξευρεθεί η καλύτερη λύση υπέρ των πολιτών. Οπότε η νομική μας επιτροπή θα έπρεπε να εμπλέκεται στον αναγκαίο βαθμό να συμμετέχει λοιπόν στην απόφαση. Καλύτερο θα ήταν το δικαστήριο να έχει δυνατότητα να εφαρμόσει τον κανονισμό του με ελαστικότητα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Χέφνα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το κοινοτικό δίκαιο αυξάνεται. Οπότε αυξάνεται και η ανάγκη για ε, δικαστήρια, για αποφάσεις δικαστηρίων. θα ήθελα να το εκφράσω ως εξή. Ναι, μεν το θέμα είναι λίγο ξηρό, αλλά είναι η πιο πολύτιμη ουσία που έχει, που, που έχει ε, δημιουργήσει η Ένωσή μας. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύουμε τους αδύνατους από επιθέσεις, από βία. Το δίκαιο ρυθμίζει τις ε, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των θεσμών, υποστηρίζει την αλληλεγγύη υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αδυνάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυστυχώς έχει όλο και μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων λόγω ακριβώς ε, της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και το Κοινοβούλιο δεν είναι κατά της αύξησης του αριθμού. Κάναμε πολύ λογικές προτάσεις για το πώς μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων και φυσικά αυτό θα βοηθούσε και τον τρόπο εργασίας του δικαστηρίου. Προτάσεις ε, έχουν κάνει ήδη συνάδελφοι. Ένα όμως είναι για μένα ακατανόητο και πρέπει να το πω σαφώς. Το Κοινοβούλιο αντιδρά στις εκκλήσεις που γίνονται, παίρνει στα σοβαρά αυτά που λένε οι δικαστές και οι πολίτες, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, προσπαθούμε και στον τριμερή διάλογο με την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Απολύτως τίποτα γιατί, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Πώς θα οριστούν οι δικαστές. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο στην κοινή μας Ευρώπη. Θα ήθελα περισσότερη ευρωπαϊκή υπευθυνότητα από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κ. Καρέμ. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο καλό βήμα για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστηρίου. Η εισαγωγή της συνθήκης της Λισαβόνας συνεισφέρει δυστυχώς στη μεγάλη καθυστέρηση και στις ορευμένες υποθέσεις που δεν έχουν ακόμα λυθεί. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης 11% επιπλέον εμπορικές διαφορές που καταλήγουν στο δικαστήριο, 37% αύξηση φορολογικών διαφορών, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για 17% επιπλέον, και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε έτσι ώστε το νομικό μας σύστημα να λειτουργήσει σωστά για να δώσουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη νομική βεβαιότητα την οποία θα πρέπει να έχουν όταν εμπορεύονται ε, διαμεθοριακά. Κάποιες πρώτες προτάσεις θα ελαφρύνουν ορισμένες καθυστερήσεις, αλλά οι προτάσεις αυτές δεν θα λύσουν δυστυχώς το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει ορισμένες φήμες που λέγουν ότι εμείς προσπαθούμε σαν Ηνωμένο Βασίλειο να μπλοκάρουμε την διαδικασία, να μην καταλήξει σε ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά εμείς με τις δικές μας νομοθετικέ εσωτερικές προτάσεις κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρος διορισμός των νέων δικαστών τον Οκτώβριο του 2012. Ο κύριος Μαστάλκα, 1,5 ε, λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Eh, eh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με τον συνάδελφο Τζέφκα τις περισσότερες φορές, αλλά όχι αυτή τη φορά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ε, συγγήτρια για τη θαυμάσια εργασία. Όπως σωστά υπόθηκε, ο αριθμός των υποθέσεων αυξάνεται συνέχεια. Αυτό έχει να κάνει με τη διεύρυνση. Σωστά λοιπόν θεωρούμε ότι στο μέλλον ο αριθμός των υποθέσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να αντιδράσουμε. Χαιρετίζω τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται μέσω της μέσω της ε, επιταχυνθής σας διαδικασίας για λήψη προσωρινών μέτρων. Και αυτή η εισαγωγή του θεσμού των αναπληρωτών δικαστών είναι αναγκαία για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Είναι δυνατότητες αυτές που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε και τη δαπάνη των δικαστικών διαδικασιών για τους διαδίκους. Γιατί όσο περισσότερο κρατάνε διαδικασίες, τόσο περισσότερα δαπανούν. Είναι σωστά λοιπόν όλα αυτά Και θεωρώ επίσης ότι είναι σωστός ο θεσμός του Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιας και εξετάζουμε τα θέματα της δικαιοσύνης υπάρχει ένα πρόβλημα σήμερα. Δυστυχώς δεν ακούγεται καλά ο Μιλκής. Ο κύριος Χέις αυτή τη στιγμή έχει προφυλακιστεί μετά από μια πρώτη ανάκριση Κρατείτε. δεν υπήρξαν μάρτυρες που να καταθέσουν υπέρ ή κατά ομιλείται λέει ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου κύριε Μπάτεν ο κύριος Μπάτεν είναι πολύ γνωστός διαμαρτυρόμενος για θέματα φορολογίας και πιστεύει ότι τα έσοδα από τη φορολογία χρησιμοποιούνται παράνομα. Ίσως σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο η κράτησή του να είναι παράνομη και ελπίζω η δημοσιοποίηση της περιπτώσεώς του να βοηθήσει. Για ένα λεπτό ο κύριος Στογιανόφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω σχετικά με την μεταρρύθμιση που προτείνεται δεν είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Ο διορισμός αναπληρωτών επιπλέον δικαστών μόνο και μόνο γιατί αρρωσταίνουν πάρα πολύ συχνά οι υπάρχοντες δικαστές είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θυμίζει την κατάχρηση εξουσίας. Γιατί αρρωσταίνουν αυτοί τόσο πολύ αυτοί μόνιμοι σχετικά με το βασικό δικαστήριο να μην ξεχνάμε ότι οι δικαστές είναι ανάμεσα στους πλέον ε, υψηλά αμοιβωμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος έχει έναν τέτοιο βουλευτή, <coughs> όχι για λόγους εθνικιστικούς, αλλά γιατί υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος να γνωρίζει το εθνικό δίκαιο και ο οποίος να συμμετέχει στο δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξουν επιπλέον αναπληρωτές δικαστές θα υπάρξει και επιπλέον επιβάρυνση των ιδίων των δικαστών. Ε, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο αριθμός εφόσον μειωθεί η αμοιβή τους έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να μην αλλάξει. Στο λόγο, στο συνάδελφο κύριο Πάουλο Ρανζέλ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται για να αναδιατυπωθεί ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο το ε, πρώτο ε, δικείο και θα ήθελα να χαιρετήσω την δημιουργία αυτής της πρότασης, την δημιουργία κανόνων για τη σύνθεση και την δυνατότητα να ανοίξει τώρα η δυνατότητα να έχουμε προσωρινούς δίκαστες σε περίπτωση κάποιου κολλήματος κάποιων δικαστών. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή η ευκαιρία μεταρρύθμισης όσον αφορά αυτό το πλαίσιο για να αυξηθεί η νομιμότητα, η δημοκρατική νομιμότητα στο δικαστήριο. Το σύστημα του κοινοτικού δικαίου, στο σύστημα του ευρωπαϊκού δικαίου, τα δικαστήρια έχουν λειτουργία να καθορίζουν προηγούμενα από νομικής πλευράς, νομολογικά, όπως το common law. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Γι' αυτό ανησυχούμε με την, ε, ε, το πρόβλημα της ε, δημοκρατικής νομιμότητας. Εφιστούμε την προσοχή σε αυτό και είναι απόλυτα αναγκαίο να αναγνωριστεί το ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Η αναφορά μιας μελέτης που πρέπει να γίνει. Αλλά σε σχέση με αυτή την πρόταση, όπως και εγώ το ανέφερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ότι όπως γίνεται στα στα δικαστήρια και στα συνταγματικά δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαιτήσουμε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις ψήφους, την ψήφιση από πλευρά των δικαστών στα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Κύριε Ραζέλ, ε, επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Αντώνιο Μασίπ Ιντάλγο. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, όπου χαιρετίζω στο πρόσωπό σας τη νέα Προεδρία, και από τους ε, μη ε, ε, δεσμευμένους τα δέσμευτα κράτη από πλευράς ε, της Κύπρου όπως ε, παλαιότερα ε, παραδοσιακά και κατά των στρατιωτικών παρεμβάσεων. Πρέπει να δραθούμε σε ευκαιρίες για μια μεταρρύθμιση του δικαστηρίου σε ευρύτερο πλαίσιο ίσως. Αλλά στόχος της Επιτροπής και του εισηγητού είναι και πρέπει να υποστηριχθεί με την ομοφωνία που έτυχε η πρόταση στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία σε σχέση με την δρομολογία που βλέπουμε ότι έχει καθυστερήσει σε σχέση με το ευρωπαϊκό ε, ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Έχει συνάδελφος κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπενόβα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπεγράμμιζε ότι το ε, δικαστήριο και το ε, πρωτοδικείο αντιμετώπιζαν υπερβολικό φόρτο εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση σε σχέση με το πλαίσιο το δικαστικό. Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς και η σημερινή δομή του ε, δικαστηρίου και να αντανακλώνται κάποιες αλλαγές που έγιναν το 2003 σαν ε, αποτέλεσμα της συνθήκης της Νίκαιας και των όσων συνέβησαν έκτοτε. 12 νέα κράτη-μέλη έχουν ενταχθεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε ότι η παραγωγικότητα έχει ναι μεν αυξηθεί από προς το δικαστηρίο όμως έχουν αυξηθεί και οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αριθμητικά. Έχει τεράστια σημασία αυτό για την χρηστή καλή λειτουργία του δικαστηρίου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια μέθοδος ε, προσδιορισμού καθορισμού των δικαστών. Ε, ζητώ από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ως ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν δηλώσεις βουλήσεως για τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και ως εκ τούτου δίνω αμέσως το λόγο στην Επίτροπο κυρία Μάλστρομ εξ ονόματος της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε φυσικά σημειώσει πολύ προσεκτικά όλες τις ε, παρατηρήσεις ε, που έγιναν σε αυτή τη συζήτηση. Μας ικανοποιεί ότι έχουμε αυτό το συμβιβασμό επί επί του οποίου συμφωνούμε χωρίς ε, να μειώνουμε τις δυσκολίες που υφίστανται στα υπόλοιπα θέματα. Θέλουμε να συνεισφέρουμε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα ο εξονόμο του Συμβουλίου, ε, ο Προεδρεύων, κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης και με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που ε, παρεμβαίνω στη συζήτηση κάτω από την δική σας Προεδρία και ελπίζω σε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Before concluding, let me just say... Ε, ε, ολοκληρώσω να πω απλά δύο λόγια για αυτό το θέμα το οποίο εθίγει για το πώς το Συμβούλιο σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα της διεύρυνσης ε, στη σύνθεση των δικαστών του δικαστηρίου. Γνωρίζετε ότι στις 20 ε, Ιουνίου η Κορεπέρ έδωσε εντολή σε σχέση με μια ομάδα από πλευρά της Προεδρίας να συνεχίσει τις σκέψεις και τον προβληματισμό για την διατύπωση προτάσεων για την επίλυση αυτού του προβλήματος μέχρι τα τέλη του έτους. Είναι κοινό στόχος και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δρομολογηθεί, να θεσπιστούν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υπερβολικού φόρτου εργασίας που έχει το δικαστήριο και με την ε, ε, νέα αυτή προσέγγιση να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και περίπλοκο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια καινοτόμο προσέγγιση, μια δημιουργική, εφάνταστη προσέγγιση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ικανοτήτων των δικαστών που θα προταθούν να αποτελούν, να συναπαρτίζουν τους, τη σύνθεση αυτού του δικαστηρίου και να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή αυτών των νέων δικαστών από κοινού με τους άλλους. Ας φανταστεί κανείς ότι θα επιλέγαμε μια ίση μέθοδο ανακύκλωσης. Ποιοι θα ανακυκλωνόντουσαν, οι 12 ή όλοι συνολικά. Όταν πρόκειται για μια χώρα θα είχε σίγουρα έναν δικαστή που θα την, θα την εκπροσωπούσε και κάποιος άλλος δικαστής άλλης χώρας θα έπρεπε να ανακυκλώνεται και η εντολή δεν θα μπορούσε να ανανεωθεί. Απλά και μόνο με αυτόν τον τρόπο συμμερίζομαι έναν προβληματισμό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να βρούμε τις πιο εύθετες λύσεις. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές από πλευράς του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή και όλους τους ευρωβουλευτές για την επικοδομητική αυτή συζήτηση για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σας διασφαλίζω ότι προσβλέπουμε στην εισαγωγή και θέσπιση νέων κανόνων και κανονισμών κατά, την, κατά το φθινόπωρο του 2012. Προσβλέπω επίσης σε επικοδομητική συνεργασία που θα συνεχιστεί από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τις προσπάθειές μας ώστε να βρούμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δικαστήριο προς όφελον όλων <clears throat> ώστε να έχουμε μια, ένα καλό ε, λειτουργούν δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κύριε Μαυρογιάννη. Και η συζήτηση ολοκληρώνεται με την παρέμβαση της ηγητρίας της κυρίας, συναδέλφου κυρίας Αλεξάνδρα Τάιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Χαίρομαι που από όλες τις πολιτικές ομάδες όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστηρίων. Η κυρία Ρέγνερ είπε ότι το πώς ακριβώς πρέπει να είναι πρέπει να συζητηθεί. Η τρίτη εξουσία πολλές φορές παραμελείται γιατί δεν μπορεί να ακουστεί αρκετά από την πολιτική. Ούτως ή άλλως η φυλακτικότητα είναι στη φύση της. Αλλά έχει ουσιώδη σημασία, το είπε και ο κύριος Χέφνα, για τους πολίτες. Και ο κύριος Κάριμ το ανέφερε, πόσο σημαντική είναι η δικαιοσύνη για τις επιχειρήσεις. Ελπίζω ότι αυτή η ομάδα φιλίας ε, που θα ε, συστήσει το Συμβούλιο δεν θα επιχειρήσει κάποιες νέες μεταρρυθμίσεις. Ε, ήδη έχει γίνει μια κάποια μεταρρύθμιση που βοήθησε να αποφασίζονται περισσότερες αποφάσεις νωρίτερα αλλά δεν θα έπρεπε να επιμείνουν να κάνουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Από ό,τι φαίνεται, ορισμένα θέματα είναι ακόμη ανοιχτά και για τα δύο θέματα και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με το δικαστήριο στο μέλλον και για τις αποκλίνουσες απόψεις που δεν τις επιθυμεί το δικαστήριο είτε αν πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά δικαστήρια. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που προέκυψαν στις συζητήσεις που ακόμη πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Αλλά υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου για τον Οκτώβριο θα υπάρξουν 17 νέοι δικαστές. Ελπίζω λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για τους επιπλέον νέους δικαστές γιατί αφορά 13 επιπλέον δικαστές το Σεπτέμβριο 2013 πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι τότε. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή κερδίσαμε κάποιο χρόνο, επειδή δεν μίλησαν διάφοροι συνάδελφοι που δεν ήταν παρόντες, να αναφέρω τις διάφορες περιπτώσεις. Οι διάφορες πολιτικές ε, ομάδες ομόφωνα μέσω ψηφίσματος αποφάσισαν ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει αυτό και λόγω ε, αλλαγής του κανονισμού. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει ε, ε, αυστηρή εναλλαγή θητιών εκεί για τους 27 ή αν θα έπρεπε ορισμένοι, έξι μόνο, να είναι από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και οι άλλοι να αντικαθίστανται. Έξι είναι ένα από τα μεγάλα κράτη και έξι από τα μικρομεσαία ε, με βάση μια εναλλαγή. Άλλη ε, λύση θα πρέπει να είναι ε, να συμπεριλαμβάνει και τον ορισμό των εισαγγελέων. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι να ορίζονται για 5-6 χρόνια κάποιοι δικαστές, Έτσι πρότεινε η Δανέζικη Προεδρία. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προτάσεις λύσεων. Το Συμβούλιο πρέπει να επιλέξει μία από αυτέ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, η εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με θέμα η κατάσταση στη Γεωργία. Ε, εξ ονόματος Αντιπροέδρου